Ε, good afternoon, all of you. Ε, Καλησπέρα. Σε όλους θα μιλήσω ελληνικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Να σας καλωσορίσω όλους στη συνεδρία μας. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους μας ομιλητές, τον δόκτωρ Στεφάν Σαλάμε, σύμβολο του Παλαιστίνου Πρωθυπουργού, και τον ε, κύριο Ροπέρτο Βάλετ από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των εε του που μας έρχονται από τη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ αντίστοιχα. Ε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, σας ενημερώνω ότι η σημερινή συνεδρία μεταδίδεται στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, και τώρα ας περάσουμε στην έγκριση του σχεδίου ημερησία διαταξή. Ε, αν δεν υπάρχουν εντηρήσει, να εγκρίνουμε την ημερησία διαταξή όπω σα έχει αποσταλεί. Περνούμε στο επόμενο θέμα, είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Ε, να πω ότι ε, σε ό,τι αφορά Κοινοβούλιο, ο πρόεδρο Ταγιάννη και ο πρόεδρο Απάς συζήτησαν πρόσφατα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρο Ταγιάννη δήλωσε ότι η στήριξη αυτή είναι αναγκαία όχι μόνο για την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της διακυβέρνησης, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο πρόεδρος Απάς εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε ότι για την οικοδόμηση μιας εύρωστης οικονομίας είναι αναγκαία η οικοδόμηση της ειρήνης. Στο τρέχον πλαίσιο ασφάλειας επανέλετε την δέσμευσή του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ισχυρή βούλησή του να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ο πρόεδρος Απάς συναντήθηκε επίση με τους πρόεδρους τους και Γιούνκερ, καθώς και με την ύπαρτη εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη. Η κυρία Μογκερίνη τόνισε ότι δεν έχει αλλάξει η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένουμε προσιλωμένοι στη λύση των δύο κρατών και την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και τη Παλαιστίνη, που αποτελεί στην προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο χαιρέτησε επίση το γεγονό ότι η ΥΠΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρο Σαπά ήρθε στο Κοινοβούλιο λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφή του Αραβικού Συνδέσμου στην Ορδανία στι 29 Μαρτίου, στο πλαίσιο τη Συνόδου Κορυφή, δόθηκε έμφαση στην επανεκκίνηση σοβαρών και αποτελεσματικών ειρευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών με βάση τη λύση των δύο κρατών και την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι ο πρόεδρος Απάς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό 23 Μαου, Κατά διάρκεια τη συνάντηση, οι Προέδρια Απά και Τραμ αναμένεται να συζητήσουν τρόπου με του οποίου θα αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία για επίτευξη λύση ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Η δική μα ευχή είναι η λύση αυτή να βρεθεί σύντομα. Ήθελα επίση να ανακοινώσω ότι η αντιπροσωπεία καταδίκασε δημόσια και απερίφραστα τον νέο οικισμό στην κατεχόμενη δυτική όχθη που ανακοίνωσε η Ισραηλική κυβέρνηση τον Μάρτιο. Επράκειτο για τον πρώτο νέο οικισμό μέσα σε 20 χρόνια και πλέον. Η νέα πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με τους οικισμούς παρουσιάζεται ως συγκρατημένη, όμως η οργάνωση Peace Now προειδοποιεί ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει το συνεχόμενο επικισμό εντός και γύρω από τους οικισμούς ακόμα και σε νέα δάφη. Μάλιστα η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να δημοσιεύσει προσκλήσεις υποβολής προσφορών για σχεδόν 2.000 καταλήμματα και να κηρύξει ως κρατικές γης σε εισαγωγικά περισσότερα εδάφη στα ενδότερα της Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, το Ισραήλ έχει μετατρέψει το 40% της Δυτικής Όχθης σε κρατικές γης από την κατοχή της δυτική Όχθης το 1967. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψει περαιτέρω οικισμού και επικισμό που θα καθιστούσαν αδύνατη τη λύση δύο κρατών. Αφού δεν θα απέμεναν επαρκή εδάφη για ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος. Εμείς εκτιμούμε τη δήλωση της ύπατη εκπροσώπους Μογκερίνη, μέσω της οποίας κάλεσε το Ισραήλ να πάψει κάθε επικιστική δραστηριότητα και αυτό που αναμένουμε είναι επιτέλους οι δηλώσεις προθέσεων να ε, μετατραπούν σε δράσεις. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει να παραμείνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στις διακρίξεις, αλλά να ακολουθήσουν πράξεις ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ενέργειες του Ισραήλ. Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη λύση και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει για να μην διαβρωθεί περαιτέρω αυτή η λύση. Σε ό,τι αφορά το ...Χάν Αλάχραμ, συνάδελφοι όπως γνωρίζετε παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τη σχεδιαζόμενη κατεδάφιση του οικισμού Βεδιούνων Χαν Ελ Αχμαρ στη ζώνη Γάμμα ε, είναι μια, ε, ένας οικισμός στο Βερίνο όπου πραγματοποιήσαμε επίσκεψη κατά τη διεύκεια της τελευταίας μας αποστολής το Φεβρουάριο στην Παλαιστίνη. Η κατεδάφιση και το 42 καταλημμάτων των οικισμών έχει προβλεφθεί για το τέλος Μαρτίου, όμως καθυστέρησε καθώς εκκρεμούσε ακόμα απάντηση του κράτους στο δικαστήριο. Στο πλαίσιο της ενεξελίξης νομικής διαδικασίας που έχει κινηθεί κατά της κατεδάφισης. Σύμφωνα με αναφορές, ο πρέσβης τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρέσβεις και των 28 κρατών μελών στο Τελαβίβ εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες κατά της κατεδάφιση αυτής, κίνηση που λέγεται ότι συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας. Οι, προσ... οι πρέσβεις δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της υποστηρίζουν από κοινού ότι η ζώνη Γ έχει κρίσιμη σημασία για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους αυτή είναι μια άποψη την οποία και εμείς συμμεριζόμαστε και μια δράση στην οποία και εμείς στηρίζουμε. αν, είχ, αν υπάρχουν εκπρόσωποι της, εξωτερικής, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης εδώ, θα ήταν καλά να μας ενημερώσουν για αυτήν τη δράση των πρέσβειων ε, σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, μπορεί να γίνει και μετά όταν θα ολοκληρώσω την ενημέρωση. Ε, σε ό,τι αφορά τη Γάζα, ως ε, αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου με την Παλαιστίνη πρώτα-πρώτα καταδικάζουμε την εκτέλεση τριών αντρών καταδικασέντος θάνατον από στρατιωτικό δικαστήριο στη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Θέλουμε να επαναλάβουμε τη σταθερή μα θέση ω κοινοβούλιο κατά τη θανατική ποινή. Επιπλέον, η Παλαιστινιακή Αρχή εφαρμόζει μορατόριο στι εκτελέσει και οι de facto αρχέ τη Γάζα πρέπει να σεβαστούν αυτή τη θέση που έχει και η Παλαιστινιακή Αρχή και να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις. Οι συνομιλίε συμφιλίωση ανάμεσα στη Χαμά και την Παλαιστινιακή Αρχή φαίνεται να έχουν επαναρχίσει. Για μας, την ευχή και ελπίδα μα, την πρωτεύουσα σημασία και ω εκ τούτου αναμένουμε από τι δύο πλευρέ να φτάσουν σε μια συμφωνία. Ε, το επόμενο θέμα που θα ήθελα να σας ενημερώσω και να κάνουμε και μια συζήτηση, να ανταλλάξουμε απόψεις, είναι για την απεργία πείνα εκ μέρου Παλαιστινίων φυλακισμένων σε Ισραηλινέ φυλακέ. Γύρω στου 1.500 Παλαιστινίων φυλακισμένων σε Ισραηλινές φυλακέ έχουν ξεκινήσει απεργία πείνα ω ένδειξη διαμαρτυρία και καταγγελία στι κακέ συνθήκε κράτηση του με την απέτηση σεβασμού στα ανθρώπινα του δικαιώματα. Η απεργία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στι 17 Απριλίου, που είναι η μέρα των φυλακισμένων, η παγκόσμια μέρα των φυλακισμένων. Δεν υπάρχει προβλεπόμενη ημερομηνία λήξη αυτή τη τόσο μεγάλη απεργία πείνα. Αποτελεί την πρώτη ευρεία κλίμακα απεργία πείνα από το Φλεβάρι του 2013, όπου 3.000 Παλαιστίνοι αρνήθηκαν τροφή για μια μέρα καταγγέλλοντας έτσι το θάνατο ενός συγκρατούμενου τους. Η παρούσα απεργία ξεκίνησε από τον ηγέτη της Φατάχ Μουρουά Μπαρκούτη, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου και ένας εκ των 13 φυλακισμένων μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου. Παλαιστίνοι από όλο το πολιτικό φάσμα συμμετέχουν σε αυτήν την απεργία μέσα από τις φυλακές εντός του Ισραήλ. Ο, ο Μπαρκούτη μαζί με όσους συγγήθηκαν της απεργίας, μεταφέρθηκα σε πλήρη απομόνωση. Μια μέρα πριν από την κήρυξη της απεργίας, ο Μαρουάν Παρκούτη κατήγγειλε στη New York Times ότι το Ισραήλ μετατρέπει βασικά δικαιώματα φυλακισμένων ε, κάτω από το διεθνή σε πρόνοια οι οποίοι μπορούν να οθούν ανάλογα με τη διάθεση των υπηρεσιών στη φυλακή και παραβιάζει όλα αυτά τα δικαιώματα. Η διεθνή Αμνηστία έχει ήδη καταγγείλει την εδώ και δεκάδε χρόνια πολιτική κράτηση Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και Γάζα σε φυλακέ μέσα στο Ισραήλ. Αποτρέπει με τον τρόπο αυτό τι επισκέψει από τι οικογένειε του φυλακισμένου. Να πράξει όχι μόνο βάναυση, αλλά κάτι που αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνού δικαίου. Το άρθρο 49 τη 4η Σύμβαση τη Γενέβη απαγορεύει ρητό τη μεταφορά φυλακισμένων από τα κατεχόμενα εδάφη σε εδάφη του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο Σύνδεσμο Παλαιστινίων Φυλακισμών αφαιρεί 6.500 Παλαιστίνου πολιτικού κρατούμενου σε φυλακέ του Ισραήλ. Ο αριθμό αυτό περιλαμβάνει 500 ε, διοικητικού πολιτικού κρατούμενου, 56 γυναίκε και 300 παιδιά. Οι φυλακισμένοι ζητούν να δοθεί ένα τέλο στη διοικητική κράτηση η οποία ουσιαστικά είναι φυλάκιση χωρίς κατηγορίες, η δίκη και θεωρείται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούν επίσης την επαλειτουργία της μηνιαίας επίσκεψης των οικογενειών τους, μεγαλύτερη σε χρόνο άδεια επίσκεψη αλλά και περισσότερα τηλέφωνα σε όλε τι φυλακέ, ώστε να επιτρέπεται επικοινωνία με του συγγενεί των φυλακισμένων. Το γεγονό ότι οι Παλαιστίνοι φυλακισμένοι κρατούνται στι φυλακέ του Ισραήλ σημαίνει ότι οι οικογένειε του πρέπει να αιτούνται αδειών οι οποίες σπανίως δίνονται, αλλά επίσης και να μπορούν να κάνουν μακρινά ταξίδια να μπορούν να δουν τους δικούς τους. Οι κανονισμοί που έχουν υπηρεσίες των φυλακών του Ισραήλ τους επιτρέπει ακόμα και να αναβάλουν προγραμματισμένη επίσκεψη οικογένεια σε φυλακισμένους επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας. Γύρω στους χίλιους φυλακισμένους έχουν αναφέρει ότι τους αρνήθηκαν να δουν την οικογένειά τους για λόγους ασφάλειας. Μπορεί να περάσουν χρόνια στη φυλακή δίχως ποτέ κανένας να μπορεί να τους δει. Πέραν αυτών, οι φυλακισμένοι καταγγέλνουν και ιατρική αμέλεια. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο Στατιστικών, από το 1967 περισσότερο από 50 Παλαιστίνοι φυλακισμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε Ισραηλινές φυλακές λόγω ιατρικής αμέλειας εκ μέρους του Ισραήλ. Οι απεργοί πείνα εφιστούν την προσοχή στι ανάγκε των γυναικών κρατουμένων για άμεσε επισκέψει από τι οικογένειε του δίχω εμπόδια και με ιδιωτική μεταφορά. Μαζί με του συμμαδέλφου μα που συμμετείχαμε πρόσφατα στην αποστολή στην Παλαιστίνη, ακούσαμε και είχαμε συζήτηση από το, με το μέλο του Παλαιστινιακού Μνομοθετικού Συμβουλίου, την Καλιδά Τζαράρ, η οποία ήταν μέχρι πρόσφατα φυλακισμένη, χωρί καμιά ε, δίκη και χωρίς ε, διοικητική διαδικασία. Ε, η Γκαλιδά Τζαράρ μας ανέφερε για τη βανασότητα με την οποία παρενοχλούνται οι φυλακισμένες γυναίκες κατά τους και όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη φυλακή κυρίως σε βάρος των γυναικών. Παλαιστίνοι φυλακισμένοι έχουν καταγγείλει τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση, τις άδικες δίκες και τις συλλήψεις και κράτηση παιδιών. Αυτό το κοινοβούλιο, μέσα από πολλά ψηφίσματα, μεταξύ άλλων και του ψηφίσματο στι 14 Μαρτίου του 2013 για την περίπτωση του Αράφατ Τζαραντάντ και την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων στι Ισραηλινέ φυλακέ, έχει ζητηθεί να εξεταστούν όλε οι καταγγελίε για βασανιστήρια και βάναυση μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων. Επαναλαμβάνουμε αυτό που ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο και στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τα αιτήματα των Παλαιστινίων κρατουμένων για συνθήκε που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω απ' όλα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Ισραήλ οφείλει να τερματίσει την παράνομη μεταφορά Παλαιστινίων κρατουμένων μακριά από την υποκατοχή Παλαιστίνη, οφείλει να σέβεται τα ανθρώπινα του δικαιώματα περιλαμβανομένου και του δικαιώματο στη δίκαιη δίκη, μακριά από βασανισμού και ταπεινωτική μεταχείριση. Οι φυλακισμένοι έχουν ανάγκη για επαρκή υγειονομική περίδαψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ανάγκη να συναντούν τι οικογένειέ του. Το κράτο του Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί όλα αυτά τα δικαιώματα. Τελειώνοντα, επιθυμώ να σημειώσω ότι οι απεργοί πείνα δεν πρέπει να υποχρεωθούν να φάνε με τη βία. Κάτι τέτοιο θα ήταν όχι μόνο ανήθικο, αλλά και μορφή βασανισμού. Ε, αυτά ως εισαγωγή αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα θα πριν να σας δώσω τον λόγο για να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και ιδιαίτερα το πώς ενεργούμε. Αλλά θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στο πρέσβη της Παλαιστίνης που βρίσκεται στην αίθουσα αν μπορεί σύντομα να συμπληρώσει κάποια στοιχεία. Ο λόγος σε εσένα κύριε πρέσβη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ως προς την απεργία πείνας για τους ε, Παλαιστίνιους κρατούμενους θα δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου και εάν μου το επιτρέψετε θα δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο του κινήματος της ΦΑΤΑΧ που βρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Όμως κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας πω ότι πολύ σωστά είπατε και πολύ ορθά αναφέρατε τα τεκτενόμενα και μετά τη συνάντηση ε, του Προέδρου ε, Αμπάς εδώ στις Βρυξέλλες στις 27 ε, Μαρτίου και μετά τις άλλες συναντήσεις που είχατε ε, έχετε λάβει πολύ μεγάλη γνώση για το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη και ορθά είπατε ότι ο πρόεδρος Αμπάς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο. Και ναι, βασιζόμαστε σε αυτή τη συνάντηση, αλλά βασιζόμαστε επίσης πάρα πολύ στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηλώσει ξεκάθαρα ότι η μόνη λύση είναι λύση δύο κρατών και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτά τα λόγια να τα τηρήσει, να μην αποκλίνει από αυτά, να διατηρηθεί η αρχή των δύο κρατών. Νομίζω ότι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμένουν σε αυτή τη λύση. Ε, όμως έχει έρθει η στιγμή να υπάρξει κάτι επιτόπου. Αυτό ζητούμε. Να αναγνωρίσουν τα 28 κράτη-μέλη το κράτος της Παλαιστίνης. Είναι το, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους μια λύση για να φτάσουμε στη λύση των δύο κρατών. Θεωρώ ότι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Έχει έρθει πλέον η στιγμή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν και το κράτος της Παλαιστίνης. Και θεωρώ ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός προς την κατεύθυνση αυτή και ο ρόλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Παλαιστίνης. Η αντιπροσωπεία σας έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και εσείς προσωπικά και σας ευχαριστώ θερμότατα για, την, ε, ε, για το έργο σας. Ανεξαρτήτως από τη συνάντηση του Προέδρου Αμπάς με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικός και απευθύνουμε έκκληση για άλλη μια φορά ε, να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να σωθεί η λύση των δύο κρατών ε, με την οποία συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αν μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στο συνάδελφο ε, για να μας μιλήσει για την απεργία πείνας και τους επικισμούς στην Παλαιστίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Το λόγο έχει ο Άντελ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ εξοχώτης, κυρίες και κύριοι, εδώ και μια εβδομάδα πάνω από χίλιους Παλαιστινίους φυλακισμένους ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν κατά της απάνθρωπης, των απανθρώπων συνθήκων κρατήσεώς τους και να προσελκύσουν την προσοχή του κόσμου σε 50 χρόνια στατιωτικής κατοχής των εδαφών της Παλαιστίνης. Πολλοί άλλοι συμμετείχαν στο κίνημα από τότε και σήμερα έχουμε, έχουμε 1500 κρατωμένους που συμμετέχουν στην όλη αυτή κίνηση. Μια απεργία πείνα δεν είναι μόνο η πιο ειρηνική μορφή αντίστασης, αλλά είναι και η τελευταία προσπάθεια για την απέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι φυλακισμένοι μας σήμερα ζητούν να τεθεί τέρμα στην απομόνωση των φυλακισμένων και στη διοικητική κράτηση. Επίσης ζητούν τη δυνατότητα να του επισκέφτονται μέλη της οικογένειας να υπάρχει ιατρική περίθαλψη και φυλακισμένοι με αναπηρία ή σε, τερματική, σε τελική φάση ασθενείας να απελευθερώνονται. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε παιδεία και πρέπει να υπάρχει επίσης, να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες όσον αφορά τη μεταφορά των φυλακισμένων και να μην υπάρχει αυτή η παρενόχληση αυτών. Έχουμε την κατοχή από το 1967. Περίπου 800.000 άνθρωποι τότε, Παλαιστίνοι τότε, έχουν φυλακιστεί από τις δυνάμεις κατοχής Είμαστε σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι έχουν απαχθεί και φυλακιστεί από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Και εγώ έχω φυλακιστεί κύριε Πρόεδρε. Περίπου 30% του πληθυσμού μας πέρασε από τις Ισραηλινές φυλακές και σήμερα το Ισραήλ έχει 6.500 Παλαιστινίους φυλακισμένους συμπεριλαμβανομένων 300 παιδιών, 65 γυναικών και 500 ανθρώπων που τελούν υποδικητική κράτηση. Η πολιτική φυλάκιση του Ισραήλ είναι παράνομη. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνέ επίπεδο και το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Σαν δύναμη κατοχή, το Ισραήλ δεν συμμορφώνεται με τι υποχρεώσει που από τη συνθήκη τη Γενέβη σχετικά με την προστασία των αμάχων υποκατοχή. Γίνεται απαγωγή Παλαιστινίων και μεταφορά αυτών σε κέντρα κράτηση στο Ισραήλ. Αυτό απαγορεύεται και είναι ανάλογο με έγκλημα πολέμου. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αγαπητά μέλη, να δει κανεί την αντίδραση των Ιζαϊνών επίκων στην απεργία πείνα. Την περασμένη εβδομάδα, άπικη, έπικη μάλλον, λοιπόν, αντέδρασαν οι έπικε στην απεργία πείνα, με αφασιστικό και βάρβαρο τρόπο. Εκατοντάδες έπικοι μαζεύτηκαν γύρω από τα στατόπεδα κράτηση για να φάνε, να κάνουν πικνίκ και να μαγειρεύσουν κρέας, ώστε να αυξηθεί το μαρτύριο των Παλαιστινίων που κάνουν απεργία πείνα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει έλλειψη λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτό εντοπίστηκε σαν μία από τι βασικέ πηγέ του ευάλωτο χαρακτήρα, ε, το του σημείου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Παλαιστινίου. Φέρει ευθύνη το Ισραήλ για την μαζική παραβίαση του διεθνού δικαίου, αναφυσβήτητα. Το διεθνέ δίκαιο απαιτεί επίση όλα τα κράτη-μέλη και μη κρατικοί φορεί να ερευνούν αποτελεσματικά τις παραβιάσεις και να διώκουν τους υπευθύνους που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου. Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι θα εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά το ανθρώπινο δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και θα πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης ότι οι όμοιροι μας στα κέντρα κράτησης του Ισραήλ αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. Επίσης καλούμε κύριε Πρόεδρε τους φίλους μας και τα μέλη εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσουν να προσθεθεί αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη επόμενη Ολομέλεια και να προσπαθήσουν επίση να συντάξουν ένα σχετικό ψήφισμα. Καλούμε το Ευρωκοινοβούλιο αμέσω να στείλει μία αποστολή για διαπίστωση γεγονότων για να ερευνήσει την κατάσταση που ισχύει όσον αφορά τι συνθήκε κράτηση Παλαιστινίων φυλακισμένων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών και τη χρήση τη διοικητική κράτηση σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 13 η Μαρτίου του 2013 υπό τις παρούς περιστάσεις θα ήταν συγκλονιστικό αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε ότι μπορεί να έχει συμβούλιο σύνδεσης με το Ισραήλ. Εναλλακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με την δύναμη κατοχής για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα παράγραφο 2 τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, και τώρα τον λόγο έχουν τα μέλη. Ξεκινώ πρώτα από τη Μάρκαρετ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, δεν είναι ε, τρομερό νέο το ότι έχουμε νιώσει τεράστια έκπληξη. Είναι συνηθισμένο νέο, γιατί είναι συνεχής οι παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Αυτό που πρέπει να ρωτήσουμε τώρα το είναι το εξή. Εάν κάποιος είναι εδώ από την υπηρεσία της κυρίας Μογκερίνη, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρει το λόγο παρακαλώ και να μας απαντήσει τι γίνεται. Τι έχει γίνει. Ναι, εντάξει, είναι απεργία πείνα, αλλά για πολύ ε, καλούς λόγους. Δεν μπορούν να συναντηθούν με τι οικογένειέ του. υφίστανται βασανιστήρια, είναι κρατούμενοι είναι μια πολύ αξιοπρεπής και ευγενής πράξη αν θέλετε. Θυμάμαι ότι το Ισραήλ ούρλιαζε σε αντίστοιχη περίπτωση για τις συνθήκες ε, κράτησης ε, μιας κρατούμενης. Τώρα με τους Παλαιστίνιους ε, κρατούμενους δεν γίνεται τίποτα. Είναι σαν να μην είναι ανθρώπινα όντα και να μην ε, τους επιτρέπεται η ανθρώπινη μεταχείριση. Επομένως, θα ήθελα πολύ καλά να ξέρω και να μάθω, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει η κυρία Μογκερίνη, τι κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα των 50 ετών κατοχής και να γίνει βασική οπτική γωνία αυτό στη συζήτηση εδώ δεν θα πρέπει μόνο να ε, ζητήσουμε να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια, να δράσουμε τώρα και να ζητήσουμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης απαντήσεις. Τι έχει κάνει, ποια βήματα έχει κάνει, η ίδια ή κάποιος άλλος ε, έχει συναντηθεί ε, με το Μαχμέτ Μπακούτι; Εμείς προσπαθήσαμε νωρίτερα, όπως θα γνωρίζετε. Το Κοινοβουλίο προσπάθησε να στείλει αντιπροσωπεία από την αντίστοιχη Επιτροπή ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλη της δικής μας αντιπροσωπείας για να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. Μας αρνήθηκαν όμως την πρόσβαση, όπως συνήθως. Και όπως συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλαλεί την κατάπληξή της στη δύσκολη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται με όλα αυτά τα ωραία λόγια, αλλά δεν γίνεται τίποτα στην πράξη. Τελικά υπονομεύουμε τους εαυτούς μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πολιτικό ε, θεσμό, εάν συνεχίσουμε να απαντούμε με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την κατάσταση που έχει τόσο πολύ χρονίσει. Και να διαμαρτυρηθούμε ότι ε, πώς το, ε, να διαμαρτυρηθούμε γιατί ο, ο, το Ισραήλ είπε ότι είναι ένα είδος τρομοκρατίας ή τρόμου αν θέλετε η απεργία πείνας και εγώ δεν νομίζω ότι αυτές οι λέξεις και αυτοί οι όροι είναι επιτρεπτές ε, στη, στη δήλωση του Ισραήλ. Άλλωστε η καταναγκαστική σύντηση είναι βασανιστήριο. θα πρέπει να θέσουμε τα σκληρά ερωτήματα στη Μογκερίνη και να, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ. Um, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε η Μαργαρέτα μόλις τώρα. Νομίζω ότι δοθέντως ότι η Καμπούτη είναι μέρος της, του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου και το ότι έχει περιγράψει αυτή την απεργία πείνας σαν τον μακρινό δρόμο των Παλαιστινίων στην ελευθερία και θεωρείται ότι είναι ο Νέλσον Μαντέλα της Παλαιστίνης. Και όπως και εσείς κύριε Πρόεδρε, όπως και η Μαργαρίτα και άλλοι, και είμαι και εγώ απογοητευμένη όσον αφορά το ρόλο που έχει διαδραματίσει ή δεν έχει διαδραματίσει η Μογκερίνη, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Ακούμε τα ίδια λόγια, τις ίδιες καταδίκες, τις ίδιες διαμαρτυρίες. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν αλλάζει όμως. Και τα αιτήματα είναι πάρα πολύ μετριοπαθή αυτών των φυλακισμένων. Και το ότι έκαναν το ίστατο βήμα να ξεκινήσουν απεργία πείνας, ξέρω προσωπικά τι κάνει αυτό στην ε, κοινότητα, στο λαό. Είχαμε δέκα φυλακισμένους που πέθαναν μέσω απεργίας πείνας στην Ιρλανδία το 1981. Το 1981. Αλλά κλείνω τα μάτια και μπορώ να σας πω τώρα που ήμουν κάθε μέρα όταν πέθανε καθένας από αυτούς τους φυλακισμένους. Τόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό. Και είναι αφάνταστο θα έλεγα δεν μπορεί να το φανταστεί κάνει, Ένα κράτο ο Παλαιστινιακό Λαό να αντιμετωπίζει 1.500 πολιτικού κρατουμένου που τελούν σε καθεστώ απεργίας πείνα. Γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό όταν διαβίας ε, δίνεται τροφή στους φυλακισμένους. Θυμάμαι τον Μάικλ Γκόχαν και τον Φρακ Στάιγ που ήταν φυλακισμένοι, που διατράφησαν υποχρεωτικά και πέθαναν λόγω καταναγκαστικής διατροφής. Είχαμε και άλλους φυλακισμένους που πέθαναν σαν αποτέλεσμα της καταναγκαστικής αυτής διατροφής. Φρίκη, απογοήτευση, ε, το είπαμε και προηγουμένως, το ξαναλέμε. Είναι σαν διάλογο κοφών. Διότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως και η Μογκερίνη κάνουν συζητήσεις, η Μαργαρίτα περισσότερο από όλου μα την στρίμωξε. Τη λέει τα ίδια και τα ίδια μα λέτε συνέχεια. Και το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε, διότι δεν υπάρχει δράση. Και γι αυτό, αυτό χρειαζόμαστε. Έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά που εφαρμόζει το Συμβούλιο. Τα σχόλια που ακούγονται. Αν ένα κράτος, μια χώρα που είναι αναγνωρισμένη, όπως είναι το Ισραήλ, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και εμπορία τιμωρητή να κινείται, θα πρέπει μέσω της υποσοπίας μας να κάνουμε κάτι περισσότερο για να το τονίσουμε. Αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Διότι είμαστε διακομματική ομάδα, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, ε, στριμώχνουμε αυτούς που πρέπει να στριμώξουμε. Αλλά λέω, στο επόμενο Στρασβούργο ίσως να είναι αργά για μερικούς από τους φυλακισμένους. Διότι κάποιοι από τους φυλακισμένους είναι ασθενείς. Και απεργία πείνας και ο αντίκτυπος της απεργίας πείνας σε κάποιους από τους κρατουμένους θα γίνει πιο αισθητό σαν αποτέλεσμα στην υγεία τους, περισσότερο από άλλους. Είμαστε στο μέσο μιας μήνης συνόδου. Θα γίνουν ψηφοφορίες την Πέμπτη. Και θα ζητούσα μέσω του Προεδρίου αυτή η αντιπροσωπεία πριν την ψηφοφορία της Πέμπτης να συναντηθούμε εκτός του ημικύκλου. Εντάξει, μόνο για να το τονίσουμε, να σταθούμε εκεί, να διαμαρτυρηθούμε, να το τονίσουμε, να φέρουμε φωτογραφίες εντός της αίθουσας, τουλάχιστον να στείλουμε ένα μήνυμα, όπως το κάναμε στην Ιρλανδία και σε όλη την Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο, να εκφράζουμε τη διεθνή αλληλεγγύη για τους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους και για το λαό, διότι αυτό που συμβαίνει είναι λάθος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουμε από τη σημερινή συνεδρίαση και ξέρω ότι, Πρόεδρε, ότι το είχατε προτείνει και πριν τη συνεδρίαση. Είπατε να κάνετε κάτι την Πέμπτη ε, πριν την ψηφοφορία και θα έλεγα αυτό να κάνουμε, να το κάνουμε σαν αντιπροσωπεία και να καλέσω και φαντάζομαι ότι μπορούμε να καλέσουμε και άλλους να έρθουν, να συμμετάσχουν απ' έξω, ώστε να προσπαθήσουμε να εκφράσουμε τη διεθνή μας αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και με τον πιο δυνατό, έτσι, έναν τρόπο που να κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρτίνα. Το λόγο ε, έχει ο ε, Μαρτίνα. Ευχαριστώ κύριε πρόταση. Συμφωνώ... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την πρόταση της ε, Μαρτίνα και με τη Μαρτίνα όταν ήταν πρόεδρος και με σένα Νεοκλή τώρα που είσαι πρόεδρος είναι σαφέστατο ότι η αντιπροσωπεία μας ε, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει το καλύτερο δυνατό για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Παλαιστίνη. Ήδη είμαι τρία χρόνια μέλος σε αυτή την αντιπροσωπεία και δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς έχουμε τα ίδια λόγια, τα ίδια παράπονα, τα ίδια προβλήματα. Και όχι δεν μιλάω για εμάς και δεν εννοώ εμάς, εννοώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μογκερίνη και τα κράτη που συνεχώς ε, επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια. Νομίζω ότι η πρόταση της Μαρτίνα μπορεί να μας κάνει να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Δεν είμαστε αποθαρρυμένοι, πρέπει να ενημερώσουμε, να σημάνουμε το καμπανάκι του συναγερμού, να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη με συνεντεύξεις τύπου, με διάφορα μέσα για να κινηθούν τα πράγματα. Και θυμάμαι έναν από τους συναδέλφους σου, νομίζω ήταν Έλληνες, δεν ήταν Κύπριος, ήταν Έλληνας, όταν, δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ Νεοκλή, σε κάθε σύνοδο της Ολομέλειας απίφθινε ερώτημα ε, στον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, τις κατα... για την κατάσταση στην οποία διαβεί ο ελληνικός λαός ε, μετά από τα αποτελέσματα των μνημονίων και της πολιτικής λιτότητας. Νομίζω ότι συνταξιοδοτήθηκε πέρσι. νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κάτι αντίστοιχο, ακόμα και δεν είναι το θέμα στην ημερήσια διάταξη, να παρεμβαίνουμε στην Ολομέλεια και να απευθύνουμε ερώτημα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην οποία διαβεί ο Παλαιστινιακός λαός. Και θα πρέπει να καλήσουμε αν θέλετε τα κράτη-μέλη να απευθυνθούμε σε αυτά. Ε, μπορεί να μην μας απαντούν, ωστόσο εδώ έχουμε μόνιμο αντιπρόσωπο κάθε χώρας μέλους να πάμε να τους δούμε τέτα τέτ, όχι με email και με τηλεφωνήματα γιατί ξέρουμε τις απαντήσεις αλλά μπορούμε να έχουμε διμελείς, τριμελείς, επιτροπές, ε, ομάδες ε, για να ε, έρθουμε σε επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο κάθε χώρα στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και να θέτουμε αυτά τα καταιγιστικά ερωτήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νεοκλή, πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Να πω ότι που παραφέρεσε ο βουλευτή είναι ο, ο πρώην βουλευτή που αποχώρησε στον ένα χρόνο, Μανώλη ο ο οποίο είναι ο άνθρωπο που κατέβασε στα 19 του χρόνια το 1941 την ναζιστική σημαία από τον Παρθενώνα από την Ακρόπολη, ο Μανώλης ο ε, τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο, διότι η αγαπητή συνάδελφος Μάρκαρετ ήταν αρκετά ε, σωστή και αυστηρή στον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, να μας απαντήσει αυτά που έθεσε και η Μάρκαρετ, αλλά θα ήθελα να αναφέρει και το ζήτημα που έθιξα προηγουμένως για την πρωτοβουλία των πρέσβες του Τελαβίβ ε, σε ό,τι αφορά τις καταφύσεις. Πού είναι ο Ευχαριστώ. Να πω ότι δεν προσεκλήθη εδώ να συμμετάσχω στη συζήτηση απλώς ως παρατηρητής. Ήρθα να ακούσω τα σχόλια. Με τα χαράς όμως να ενημερώσω την ιεραρχία μου για τα σχόλια που ακούστηκαν από τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Όμως, εφόσον έχω το λόγο, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Προφανώς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εξεφράστησαν προηγουμένως για την μοίρα των απεργών πείνας στις Ισραηλινές φυλακές. Νομίζω ότι είναι σαφέστατο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα θεσμικά όργανα. Στο σύνολό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφέστατη πολιτική, υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, βάσει των αρχών της λογοδοσίας, που είναι ακρογωνίως λήθος για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και έχετε πολλά συμπεράσματα του Συμβουλίου που επανεπιβεβαιώνουν αυτές τις αρχές. Επίσης θα μπορούσα να αναφέρω ότι έχουμε αρκετούς αξιωματόχους της ιεραρχίας που έδρασαν με διακριτικότητα πίσω από κλεισμένε πόρτες, ούτω ώστε να θέσουν το θέμα των απεργών πείνας. Δεν ξέρω αν συγκεκριμένη περίπτωση έγινε αυτό, ξέρω άλλες περιπτώσεις όμως όπου αξιωματούχοι έδρασαν σε παρόμοια κατάσταση. Ακούστηκε ένα άλλο σχόλιο αφορούσε τον κανάλ, το κανάλ Αλμάρ, την ε, κοινότητα των Βεδουίνων που κινδυνεύει να κατεδαφιστεί. Να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδρασαν με στεναρότητα για την υπεράσπιση αυτής της κοινότητας που είναι κοντά στο Ιουάν σε πολύ στρατηγική τοποθεσία για το μέλλον της λύσεως των δύο κρατών έγιναν δημόσιες δηλώσεις επιτόπια από αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών, έγιναν διπλωματικής φύσεως επισκέψεις, ε, η, εξωτερική, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης κατέβαλε διπλωματικές προσπάθειες, συνέβαλε σε μια έκθεση που συνέταξε η Wall Street Journal για τη μοίρα της κοινότητας, επιπλέον, όπως ανέφεραν και τα ΜΜΕ, επικεφαλής αντιπροσωπείας στο Τελαβίβ, μαζί με εκπροσώπους των 28 κρατών μελών, έδωσαν σαφέστατο μήνυμα προς τις Ισραηλινές αρχές. Δεν μπορώ παρά να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε καταλήψει κανένα μονοπάτι, χρησιμοποίησαμε κάθε δυνατότητα στα θεσμικά όνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να επερασπιστούμε επιτόπου αυτή την κοινότητα. Επίσης, ένα ιδιωτική σφίστο σχόλιο, αν με επιτρέπετε, δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι, να κατηγορεί κανεί διάφορα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το κάτω-κάτω μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά μόνο αν δρούμε από κοινού. Και έχουμε κοινέ ανησυχίε και έχουμε κοινού στόχου. Άρα απευθύνω έκκληση προ όλου. Συνεργαστείτε μαζί μα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πραγματικά και δυσχερέστατα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι και κάποιοι Ισραηλινοί εκεί επί τόπου. Αλλά θα επιβάσω τα μηνύματα και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ε, Όμω είμαι αναγκασμένο να κάνω ένα σχόλιο. Ε, είναι ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Και ο ρόλο του Κοινοβουλίου είναι ελέγχει και ενίοτε εκεί που θεωρούμε ότι δεν προχωράει σωστά ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ασκούμε την κριτική, να ασκούμε τον έλεγχο. Ε, θεωρώ ότι αυτό που προβάλλουν τα μέλη της αντιπροσωπείας και το Κοινοβούλιο τις περισσότερες φορές είναι οι θέσεις αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να ακολουθεί. Και όπου υπάρχει, κατά την άποψή μας, αδράνεια, εμείς οφείλουμε αυτό να το κριτικάρουμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι ούτε η Επιτροπή, ούτε καμιά υπηρεσία θα πρέπει να νιώθει ότι επειδή ασκούμε αυτή την κριτική ότι θέλουμε να είμαστε σε μια σύγκρουση. Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε όλοι είναι επιτέλου, αυτό που ανάφεραν και άλλοι συναδέλφοι, το είπα και εγώ στην εισήγηση μου, να περάσουμε από τα λόγια στι πράξεις. Να περάσουμε από τι διακηρύξεις στι δράσει για, για όλα αυτά τα εγκλήματα ε, που γίνονται στην Παλαιστίνη ε, και όλοι τα βλέπουμε και όλοι τα συναντούμε. Ε, πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να δώσω τον λόγο πολύ σύντομα στον εκπρόσωπο ε, της ΦΑΤΑΧ για να μας μεταφέρει δύο μηνύματα και μετά θα δώσω τον λόγο στην... Ε, έχουμε μαζί μας ε, μια μη κυβερνητική οργάνωση, είναι τη Solidarité Palestine, να μας πει και αυτή δύο λόγια. Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον εκπρόσωπο της ΦΑΤΑΧ να είναι πολύ σύντομος. Ο λόγος σε σένα, Thanks, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μας τους φίλους εδώ που υποστηρίζουν το αίτημά μας και την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους απεργούς πείνας. Σήμερα είμαστε εδώ για να στείλουμε δύο μηνύματα. Ένα πρώτο μήνυμα από τον Μαρουάν Μπαργούτη, τον επικεφαλής της απεργίας πείνας και το δεύτερο μήνυμα, το μήνυμα από το κίνημα της ΦΑΤΑΧ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, το λόγο τώρα έχει η Σιλουά, είναι εκπρόσωπος της ε, Solidarité Palestine εδώ στο Βέλγιο. Ναι, Σιλουά. Hello, thank you very much. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που δώσατε περιθώριο να συζητηθεί αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Συμμετείχα σε μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα τους απεργούς πίνεας και η έκθεση φωτογραφίας ταξίδεψε και στην Παλαιστινή και τα μέλη των οικογενειών των απεργών πίνας συγκινήθηκαν ιδιαίτερως με το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά έχουν ήδη υποθεί, δεν θα επανέλθω. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξής. Πολλά από τα αιτήματα των απεργών πείνας έχουν να κάνουν με δικαιώματα που τους ε, καταργήθηκαν. Δηλαδή πρέπει να ξαναπαλέψουν ε, για να ξανακερδίσουν πολύ βασικά δικαιώματα τα οποία στερήθηκαν. Για παράδειγμα το δικαίωμα να πιάσουν το χέρι ε, κάποιου που τους επισκέπτεται. Το δικαίωμα στη βασική ιατρική περιθέλψη. Στις συνθήκες μεταγωγών μεταφοράς για τους ασθενείς τιμωρούνται οι κρατούμενοι για τις πράξεις τους, για το ότι μιλούν ανοιχτά, για το ότι ζητούν αλληλεγγύη και ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Τους πήραν το αλάτι που είναι πολύ βασικό για τους ηλεκτρολίτες και για τη ζωή τους. Τους πήραν ε, τα μπουκάλια νερού, άρα πρέπει να σηκωθούν και να περπατήσουν μέχρι τη βρύση για να πιούν, κάτι το οποίο τους εξαντλεί. Και αυτό είναι τιμωρία. Ουσιαστικά είναι όλα αυτά τιμωρίε για να σταματήσουν την απεργία πίκινας. Όλο και περισσότεροι μπαίνουν στην απομόνηση, δεν υπάρχουν επισκέψεις, ούτε καν επισκέψει από τους δικηγόρους τους. Ε, δίνουν αγώνα για να κερδίσουν το δικαίωμα να δουν τους δικηγόρους τους όταν κάνουν απεργία πείνας. Και όταν οι δικηγόροι πήγαν στη φυλακή ακυρώθηκε η επίσκεψη γιατί σήμανε συνεγερμό και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συνεγερμού. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ βασικά τα αιτήματα, πάρα πολλά έχουν να κάνουν με, την, με το να έχουν δικαιώματα που είχαν στο παρελθόν και του τα ε, κατήργησαν. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν ικανοποίηση στα αιτήματά τους. Η ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων είναι ε, το βασικό, είναι ο πυρήνας και οφείλουμε ε, να το επιτύχουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα. Όταν ο Υπουργό τη Δημόσια Ασφάλεια είναι και επικεφαλή του σοφρονιστικού συστήματο του Ισραήλ και είναι εταίρο και λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα, για σχέδια επενδύσεων σε ανακριτικά και τεχνικές. Αυτό υπάρχει στο project Ορίζοντας 2020. Όταν έχουμε άμεση εταιρική σχέση, δηλαδή με ανθρώπους που καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε και μέσα πίεση να ασκήσουμε ε, ε, προς αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν αμφισβητήσουμε το ότι είναι εταίροι μας, γιατί ξανά και ξανά επανειλημμένος έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε εταίρους στο Ισραήλ γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε το διάλογο μου ανοιχτό. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχουμε εταίρους στο Ισραήλ για να μπορούμε να ασκούμε πίεση. Ε, τότε ας χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σημαντικές της σχέσεις για να ασκήσει αυτή την πίεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε το Ισραήλ να ε, να είναι μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν, είναι, δεν αποτελούν ε, μέρος του καταλόγου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να ολοκληρώσει για να μπορεί να έχει εταιρική σχέση με κάποιον δυστυχώς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ε, αρθρώσουμε το λόγο μας και να ασκήσουμε πίεση για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες. Οι συναδέλφοι μου είναι αυτά που επαναλαμβάνουμε κατά κόρο και εδώ στις συνεδριάσεις μας αλλά και στις Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ε, να μου επιτρέψετε ε, πολύ σύντομα να διαβάσω το μήνυμα που μας ε, έχουν δώσει οι συνάδελφοι που τη φαντάγει εκ μέρους του Μουρουάν Μπαρκούτη είναι μια επιστολή που βγαίνει μέσα από το κελί τη απομόνωση και απευθύνεται ε, σε όλους τους αδερφούς. To our friends throughout the world. am Φίλους στον κόσμο, σας μιλώ σήμερα και μιλώ για το, από το μικρό μου κελί της απομόνωσης. Στο επίκεντρο χιλιάδων φυλακισμένων και εκφράζω την άποψη των φυλακισμένων. Και αποφασίσαμε με τις χιλιάδες φυλακισμένους να πολεμήσουμε τη μάχη της ελευθερίας εξωπρέπειας. Τη μάχη της τιμής και του ηρωισμού. Τη μάχη της απεργίας πείνας για να περιστηθούμε το δικαίωμά μας στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Θα κάνουμε αυτή την απεργία για να αντιπαταχθούμε στη συνεχή βίαιη πολιτική ε, κατοχής, απαγωγής, βασανισμού, ιατρικής αμέλειας, αυθαίρετης τιμωρητικής αντιμετώπισης των φυλακισμένων και των οικογενειών τους, στερώντας τους από το δικαίωμα πρόσβασης. Επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας για την απεργία πείνας, ανεξάρτητα θυσιών, ανεξάρτητα πόνου και μαρτυρίων. Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτό το λαό και είμαστε σε θέση να έχουμε σταθερή θέση, να αντισταθούμε μέχρι ότου να αποκτήσουμε δικαιώματά μας που εγγυώνται ο νόμος και οι διεθνείς συμβάσεις. Αυτές οι μάχες συμπίπτουν με την ημέρα των Παλαιστινίων φυλακισμένων. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνοι υπήρξαν θύματα αυθερέτων συλλήψεων, φυσικών και ψυχολογικών βασανιστήριων και ταπείνωσης κάθε είδους από πλευράς δυνάμων κατοχής. Ο αδελφός σας Μουρουάν Παρκούτ. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, διότι έχουμε εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη. Θα σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι ε, πρώτα πρώτα εκ μέρους της αντιπροσωπείας θα εκδοθεί σήμερα ανακοίνωση τύπου αναφορικά με το ζήτημα των Παλαιστινίων κρατουμένων ε, μετά από τη συνάντησή μας. Για να εκφράσουμε ακριβώς την καταδίκη μας και τις δικές μας απόψεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ε, το έθεσε και εδώ η, η Μαρτίνα. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η πρόταση την Πέπτη πριν από τις ψηφοφορίες που θα είναι μαζεμένη και ολομένα του Κοινοβουλίου έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας να, κάνουμε μια, ε, να προβάλλουμε το αίτημα του Πασέρε. Μια εκδήλωση συμβολική διαμαρτυρίας για να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Και το τρίτο, βεβαίω αυτά που έχει προτείνει ο Άντελ από την Πρεσβεία της Παλαιστίνης, ε, θα εξετάσουμε ενδεχομένως σε δύο εβδομάδες όταν θα έχουμε την Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Έχει δίκιο η Μαρτίνα, δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί. Ε, πρώτα πρώτα το θέμα εάν μπορούμε να προτείνουμε ψήφισμα ε, στην... Επίσης να κάνουμε αυτό που πρότεινα για την αποστολή. Θα, θα προτείνουμε για ψήφισμα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και να εξετάσουμε τη δυνατότητα ε, επίσκεψης αντιπροσωπείας για να δει επιτόπου την κατάσταση των φυλακισμένων. Ε, αλλά αντιλαμβάνεστε επειδή αφορά το Ισραήλ πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου, ε, το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ε, για να υπάρχει επίσκεψη, για να δούμε επιτόπου στην κατάσταση με τους απεργούς πείρας και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αυτά είναι τα βήματα που θα προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα γύρω από αυτό το θέμα. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα να μου να, να περάσω, να δώσω τον λόγο ε, στους καλεσμένους μας για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων γύρω από σχετικά με την Παλαιστινιακή Αθεκτικότητα. Ε, έχω μπει κι άλλες ε, που είναι στην ατζέντα μας, τους φιλοξενούμενους μας, να πω ότι ε, πραγματικά εδώ στο Κοινοβούλιο πολλές φορές συζητήσαμε τη στρατηγική συνεργασία της Ευρωπαϊκής με την Παλαιστίνη, και την ανάγκη να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεδηλωμένο πολιτικό στόλο για τη στήριξη των δύο κρατών. Βεβαίω, για να μπορεί η Παλαιστίνη να λειτουργήσει ω πραγματικό κράτο, ε, πρέπει, ε, ε, πρέπει να συνεχιστεί η πορεία προόδου τη για την επίτευξη τη πολιτική υπόσταση. Απαιτείται πρώτα πολιτική βούληση. Εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο έχουμε κάνει το μέρο που μα αναλογεί με την Πρώτα πρώτα με την αλλαγή του ονόματο τη Παλαιστινιακή Αρχή, αυτό που καλέσαμε πάρα πολλέ φορέ τα κράτη-μέλη, είναι να προχωρήσει η αναγνώριση τη Παλαιστίνη ω ε, Παλαιστινιακού κράτου. Ε, γι' αυτό πρέπει να σα πω, υποδεχόμαστε σήμερα του ε, προσκεκλημένου μα επισκέπτε, προκειμένου να εξετάσουμε τρόπου τη ε, αντιμετώπιση τη κατάσταση, ενίσχυση τη ρόλη του Παλαιστινιακού λαού να ξεπερνά όλο έναντι χειρέστερη κατάσταση, ένα πλαίσιο παλαιστινιακής ανθεκτικότητας, το οποίο να σας πω ότι για πρώτη φορά συζητούμε αυτό το θέμα εδώ ε, στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα καλέσω πρώτα τον δόκτωρ Στεφάν Σαλάμε, ε, σύμφωνο της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, ο οποίος έχει ηγηθεί της ομάδας σχεδιασμού υπεύθυνη για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής Παλαιστίνης και τομεακής στρατηγικής ε, ο 2017-2022, ο Δ. Σαλάμι θα μα ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα διάφορα Υπουργεία τη Παλαιστινιακής Αρχή για την αντιμετώπιση τη κατάσταση και για ενίσχυση του Παλαιστινιακού λαού. Έχει τον λόγο ο Δ. Ε, Στεφάν Σαλάμι ε, για 10 λεπτά. Ο λόγος σε σένα, Δ. Στεφάν. Καλησπέρα, αξιότιμη κύριε Νεοκλήση Σιλικιώτη, πρόεδρε της αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Παλαιστίνη, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, μέλη της αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, εξοχότητά σα, κύριε πρέσβη Αλφάρο, πρεσβευτή της Παλαιστίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βέλιο και το Λουξεμβούργο, κύριε Ρομπέρτο Βάλενς, εκπρόσωπο του ΟΗΕ στην Παλαιστίνη, Αλμανσούρ Μπανφάτα, διευθυντή του τμήματος καταπιστεύματος της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Κυρίε και κύριοι, είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και να μιλήσω για την αντοχή των Παλαιστινίων. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά αισθάνομαι ταπεινότητα έναντι των δηλώσεων που ακούστηκαν σήμερα από τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου κυρίως αυτά που υπόθηκαν για την κατάσταση των φυλακισμένων μας. Οι φυλακισμένοι μας είναι απόδειξη, υπόδειγμα σταθερότητας και ανθεκτικότητας Παλαιστινίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθική ευθύνη συνεπώς να δράσει για να προστατεύσει και να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως τα δικαιώματα των Παλαιστινίων φυλακισμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία της με ένα κράτος που συνεχώς και σκοπίμως παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Παλαιστίνη υποφέραμε από την κατοχή την Ζαλινή επί 50 χρόνια τώρα. Ο αποκλεισμό της Γάζας συνεχίζεται τώρα για πάνω από μια δεκαετία. 100 χρόνια από την δήλωση του Μπελφόρ και 69 χρόνια πέρασαν από την Άκβα. Οι Παλαιστίνοι αντιστέκονται κατά των ξένων επικοινωνικών δυνάμεων επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε πτυχή της ζωής μας, της ζωής μας ως Παλαιστινίων, περιορίστηκε σε όλους τους τομείς της. Η δυνατότητά μας εργαστούμε, Φερρυπίν, να ταξιδέψουμε, να ζήσουμε, να παράξουμε, να εμπορευτούμε και να διχειριστούμε τις υποθέσεις μας. Όλα έχουν επηρεαστεί. Εμείς παρατηρούσαμε, βλέποντας τη χώρα μας και την πατρίδα μας να κατακαιρματίζεται όλο και περισσότερο. Και έχουμε μείνει με όλο και λιγότερα πράγματα. Αλλά ως Παλαιστίνοι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανθεκτικοί. Το αποδείξαμε αυτό επανειλημμένα τα τελευταία 100 χρόνια με το δικό μας τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη τους επιβληθέντες περιορισμούς από τις δυνάμεις κατοχής στην Παλαιστίνη, είχαμε αξιέπαινη πρόοδο ανάπτυξης. Είμαστε μια χώρα μέσου, χαμηλό, εμέσου επίπεδου με πολύ καλά επίπεδα όσον αφορά την εκπαίδευση των γυναικών υπόδειγμα στον αραβικό κόσμο. Παρά τα αυτά ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα ανθρωπιστικής φύσης και αναπτυξιακές ανάγκες λόγω της Ισραηλινής κατοχής. Η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επιμακρών. Καθημερινά βλέπουμε η γη μας να κλέπτεται να αρπάζεται από παράνομους επικισμούς των Ισραηλινών. Βλέπουμε τα σπίτια του λαού μας να κατεδαφίζονται ή να καταλαμβάνονται και παιδιά 12 χρονών, τόσο νέα συναμβάνονται, απάγονται, φυλακίζονται στο, και πηγαίνουν στο Ισραήλ. Πέρσι, ε, για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το UNDP, καταφέραμε να συγκαλέσουμε την πρώτη διάσκεψη στην αντοχή της Παλαιστίνης. Πιστεύουμε ότι είναι και η ώρα να αλλάξει ο τρόπος χορηγήσεως ενίσχυσης προς την Παλαιστίνη. Η διάσκεψη μας υπενθύμησε ότι η παλαιστινιακή αυτή αντίσταση, η αντοχή διαβρώνεται και θα πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου. Η αντοχή είναι ένα φύγημα στήριξης, απελευθέρωσης και χειραφέτησης, αλλά μόνο υπό τη μεταμορφωτική της μορφή. Σαν κυβέρνηση έχουμε διατυπώσει ένα νέο τρόπο αυτής της μεταμορφωτικής αντοχής. Δεν είναι κάτι που αφορά την επιβίωση, την αναταραχή της κατοχής, αλλά να περάσουμε πιο πέρα, να μεταμορφωθούμε και να ξαναποκτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Αυτό είναι θεν για κάποιους λαούς, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το λαό που τελεί κατοχή, όπως είναι η Παλαιστίνη. Η εθνική μας πολιτική έχει ένα θεματολόγιο. Στηρίζεται σε αυτά τα ιδεώδη της αντοχής που σας περιέγραψα. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε όλους τους Παλαιστινίους. Επί σειρά ετών ακούγαμε τη νέα ιδέα της αντοχής. Αντοχή είναι η ιδέα να αντιμετωπίζει κανείς τα προβλήματα της κρίσης και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις τραυματικής φύσεως. Όμως δεν θα πρέπει που να γίνει ένα άλλο σύνθημα που θα είναι κενό περιεχομένου. Χρειάζεται πρακτικές προσεγγίσεις. Χρειάζεται εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι βασικοί κινδυνοί, οι πιο μεγάλοι όπως η κατοχή, η βία, η ανασφάλεια της διατροφής, η αδικία και άλλα προβλήματα. Ως Παλαιστίνοι όμως είμαστε ήδη ανθεκτικοί. Έχουμε εφαρμόσει την αντοχή μέσω της δικής μας εγενούς ε, ενίας της Σομότς επί χρόνια, επί δεκαετίες. Η ύπαρξή μας, η επιμονή μας, η αποφασιστικότητά μας έχουν αποδείξει ότι έχουμε αντοχές. Μετά την Ισραηλινή κατοχή το 1967 οι Παλαιστίνοι εφάρμοσαν το σουμούντ, η σταθερότητα, η αντοχή, οπω το λέμε. Ε, και υπάρχουν πολλοί τρόποι σουμούντ. Βλέπουμε Παλαιστίνοι που δεν έφυγαν από το χώρο του ακόμα και όταν αντιμετώπισαν βίες επιθέσει, Μία μορφή σουμούντ. Βλέπουμε τον Γεωργό που ξαναφυτεύει Παλαιστινιακέ ελιέ, ανεξάρτητα από τι φορέ που καταστρέφονται οι ελιές. Βλέπουμε την οικογένεια που μένει στα σπίτια τη, αντιμετωπίζοντας και τις μπουλντόζες ακόμα τα, τα παιδιά της Παλαιστίνης που περπατούν χιλιόμετρα ολόκληρα στο δρόμο, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη βροχή για να πάνε στο σχολείο. Θυμάμαι το 1988 όταν ο Ισραηλινός στρατός έκλεισε το Πανεπιστήμιο του Μπιλζάιτ για τρία χρόνια. Οι Παλαιστίνοι πήγαιναν και παρακολουθούσαν μαθήματα στα σπίτια και κάθε φορά συλλαμβανόταν όταν τους βλέπαν να κουβαλάνε βιβλία για να πάνε στα σπίτια για να μελετήσουν και για να μάθουν. Οι Παλαιστίνοι έχουν πολλά να προσφέρουν όσον αφορά την έννοια τη αντοχής. Μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα πώς το εκπαιδευτικό σύστημα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί κατά από τις επιθέσεις και την κατοχή και τι επιθέσει των Ιζαρινών αρχών. Πώς η περίθαλψη η τομέα τη υγεία μπορεί να συνεχίζεται σε τέτοιες παρόμοιε περιστάσει. Το Σουμούντ παραμένει κοντά στην καρδιά μας, στην καρδιά των Παλαιστινίων. Στις παρεμβάσεις μας, σε σύμπραξη με τη διεθνή κοινότητα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ριζικά αίτια της Παλαιστινιακής καταστάσεως. Πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε όχι βραχυπρόθεσμη βοήθεια που ε, θεραπεύει μόνο τα συμπτώματα και όχι τα αίτια. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντοχής και μέσω της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας είναι μια καλή αφετηρία. Αναφέρεται στην αντοχή, ποικιλοτρόπος, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακή βοήθεια, μείωση καταστροφών, προβλημάτων αλλαγής του κλίματος, προσαρμογής, αποφυγής συγκρούσεων και ειρήνευση. Αλλά πολύ λίγες αυτές τις πολιτικές άμεσα σχετίζονται με την κατάσταση που επικρατεί και την αντοχή των Παλαιστινίων, διότι επουδενή δεν αναφέρεται στην κατοχή Όμω η έννοια τη αντοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση αναδύεται σταδιακά το 2007 για να αντιμετωπιστούν οι εξελίξει εκεί, οι συγκρούσει με οριστικό τρόπο. όμω, αυτό που μα αφορά περισσότερο από όλα αυτά, εμά του Παλαιστινίου, είναι το σχέδιο δράση του 2013 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντοχή σε χώρε που αντιμετωπίζουν κρίση για την περίοδο 2013-2020. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ριζικά αίτια των κρίσεων και των συγκρούσεων, ενισχύοντας εθνική, τοπική δυνατότητα αντοχής, παρουσιάζοντας εργαλεία για την υποστήριξη αντοχής, όπως το ΣΕΡ και το NGIR, όμως η Παλαιστίνη δεν συμπεριλαμβάνεται σε κανένα από τα καταπιστεύματα, trust funds, για την αντοχή που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα θέλαμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει και την Παλαιστίνη στην πολιτική της για την υποστήριξη της εντοχής στις αφρικανικές χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι δεν συμπεριλαμβάνεται για την ώρα η Παλαιστίνη. Η νέα, το νέο μας θεματολόγιο που διαμορφώθηκε εδράζεται και επί τη μεταμορφωτική, μετασχηματιστικής αντοχή. Έχουμε εθνικό θεματολόγιο πολιτικών και έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, προσέγγιση και σχεδιασμό και ελπίζουμε να αντιμετωπιστούν έτσι τα ριζικά αίτια των προβλημάτων μα που αντιμετωπίζουμε ω Παλαιστίνοι. Μέσω αυτού έχουμε τρει βασικού πυλώνε εθνικέ προτεραιότητε, διεθνεί πολιτικέ και 115 πολιτικέ παρέμβασεις που γνωρίζουμε ότι θα μα βοηθήσουν να πετύχουμε του στόχου μα. Το μονοπάτι προς ανεξαρτησία μέσω του τερματισμού της κατοχής, η επίτευξη της ανεξαρτησίας και η δημιουργία της εθνικής ενότητας. Δεύτερος πυλώνας αναφέρεται σε κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και καλύτερες υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες. Εκεί θα εξασφαλίζουμε το ότι θα είμαστε θα ακολουθούν πολιτική που εδράζεται των πολιτών και θα είναι διαφάνεια, ε, θα εφαρμόζεται διαφάνεια από την κυβέρνηση, βιώσιμη ανάπτυξη των τύπων πυλώνα. Όλο ο λαό θα πρέπει να είναι έτοιμο για το μελλοντικό μα κράτο. Δεν θα έχουμε ανασφάλεια διατροφή, δεν θα έχουμε φτωχά νοικοκυριά, θα υπάρχει παιδεία για όλου, περίθαλψη για όλου, εξωπρεπή εργασία για όλου και θα υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη και οι νέοι και οι γυναίκες θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν του μέλλοντό μα ω Παλαιστίνοι. Όλοι μαζί αυτοί τι πυλώνε μπορούν να βοηθήσουν να αναπτυχθεί η αντοχή των Παλαιστινίων και των κοινοτήτων, ξεκινώντα με το Εθνικό Θεματολόγιο Πολιτική. Στη διάσκεψη της αντοχής που διοργανώθηκε πέρσι φτάσαμε στην ομάδα κρούσης για την αντοχή που διαμορφώθηκε που είναι αποτέλεσμα της ε, και έχουμε το Γραφείο Συντονισμού, έχουμε μια υπηρεσία ανοικοδόμησης της Γάζας και με όλα αυτά αναζωογονούμε την αντίσταση των Παλαιστινίων, την αντοχή των Παλαιστινίων. Πιστεύουμε ένθερμα στη μετασχηματιστική αντοχή μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Είναι ένα μέσο που βοηθά να μεταμορφώσει το, το σύστημα ενισχύσεων από τις παρούσες δομές που τεχνικά ε, κατανέμουν τις διάφορες πανεμβάσεις και τη βοήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο όπως και το Παλαιστινιακό, αντιμετωπίζουμε καταστροφικές κρίσεις μαζί με τα αναπτυξιακά προβλήματα και χρειάζεται και είναι κρισίμου σημασία μια νέα προσέγγιση. Η μεταμορφωτική αυτή αντοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντάξει και τις δύο διαστάσεις. Απλή ανθρωπιστική βοήθεια δεν αρκεί, βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι δυνατή υποκατοχή, οπότε η αντοχή είναι ο σωστός δρόμος. Αντοχή είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Να έχουμε ενοποιημένο σαφή στόχο και ένα πλαίσιο για να προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο στόχο. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επαγρυπνεί, να εξασφαλίζει ότι οι παλαιστινικές φωνές θα εισακούγονται όταν σχεδιάζονται νέα προγράμματα. Θα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες του λαού, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία θα πρέπει και να αντιμετωπίζονται και τα διάφορα προβλήματα στον δρόμο προς την επιτυχία. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται η ενίσχυση, να γίνει αποτελεσματικότερη, να λάβει υπόψη ανάγκη κοινότητα και να έχει νόημα για του Παλαιστινίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργασία, μέσω κοινών δράσεων, μέσω στρατηγικών επαφών, μέσω συμπράξεων, μέσω του συντονισμού μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικού τομέα και τη διεθνού κοινότητα ε, ενισχύσεων. Μετά τη διάσκεψη αντοχής των Παλαιστινίων που έλαβε χώρα το 2016, έχω με βρει νέε συμπράξει και συνεργασίε και δίκτυα μεταξύ ανθρωπιστικών και αντισιακών φορέων και όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ριζικά αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι. Σαν κυβέρνηση μέσω του γραφείου του Πρωθυπουργού έχουμε δείξει ότι είμαστε αφοσιωμένοι στην αντοχή, δημιουργώντας την Task Force για την αντοχή των Παλαιστινίων. Αυτή η ομάδα κρούση έχει σε εκπροσώπηση από όλου του εμπλεκόμενου φορεί και παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε καθαρό οδικό χάρτη για το μέλλον και συντονισμένο πλαίσιο για να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Μαζί δημιουργούμε μια, ένα κονσόρτσιουμ αντοχής με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Ακούμε τις απόψεις τους για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για να αυξήσουμε την αντοχή των Παλαιστινίων. Ήρθε η ώρα για την αλλαγή για την Παλαιστινή. Ήρθε η ώρα αυτή. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων σας για να συμβούν αυτά. Εάν όχι τώρα, τότε πότε. Αν όχι εμείς, τότε ποιος. Κινητοποιώντας την έννοια της μετασχηματιστικής αυτής αντοχής, μπορούμε να καταστήσουμε δυνατή την αλλαγή για να βελτιώσουμε τη ζωή των Παλαιστινίων, να τεθεί τέρμα στην κατοχή και τελικά να πετύχουμε την εξαρτησία της Παλαιστίνης και την αυτοδιάθεσή της. Ήρθε η ώρα να τερματιστεί μία από τις μεγαλύτερες ε, δυνάμεις απεικιοκρατίας στον κόσμο και να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Σαν κυβέρνηση είμαστε έτοιμοι για κυριαρχία. Θέλουμε να βρούμε μια νέα λύση σε ένα παλιό πρόβλημα. Θα πρέπει να καινοτομήσουμε και να ξεπεράσουμε τις ισχύουσες παρεμβάσεις. Θα πρέπει να απελευθερώσουμε την Παλαιστίνη από την κατοχή και να κατασκευάσουμε βιώσιμη, βιώσιμη, ενωμένη Παλαιστινιακή, Παλαιστινιακό κράτος η καθεστική ατάξη στο παρόν status quo δεν λειτουργεί. Βρήκαμε μια νέα λύση για να αλλάξει η καθεστική ατάξη στην Παλαιστίνη. Χρειαζόμαστε τη δική σα στήριξη και τη στήριξη διεθνού κοινότητα, ώστε όλα αυτά να συμβούν. Και επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όταν μιλούμε για παλαιστινιακή αντοχή, δεν αναφερόμαστε μόνο στην αντοχή για επιβίωση. Εννοούμε παλαιστινιακή αντοχή για απελευθέρωση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αντοχής για επιβίωση και αντοχής για απελευθέρωση. Η αντοχή για μας είναι κάτι συλλογικό, συλλογική πράξη συνειδητή για να αντιμετωπίσουμε τη βία, την κατοχή, την αδικία, την ανασφάλεια και όλα τα είδη των κινδύνων. Και βασιζόμαστε στη συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ώστε αυτή να δράσει και να μας υποστηρίξει στο μονοπάτι μας προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Τελικά, δεν χρειάζεται να επενθυμίσω σε όλους σας ότι η λύση των δύο κρατών είναι ευρωπαϊκή ιδέα, η οποία εισήχθη το 1980. Δεν χρειάζεται να πω ότι η λύση των δύο κρατών κινδυνεύει. Αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο. Συστηματικά το Ισραήλ καταστρέφει κάθε ελπίδα για υλοποίηση της λύσεως των δύο κρατών. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθική ευθύνη να δράσει, να προστατεύσει τη λύση των δύο κρατών και να εξασφαλίσει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όπως σωστά είπε και ο προσβευτής μας στην αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ένα από τα δύο κράτη. Ένας τρόπος να προστατευτεί η λύση των δύο κρατών είναι αμέσως τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη και να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε και να καλέσω ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί και να θέσει άμεσα αυτά τα ζητήματα όταν μιλάμε για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να συνδέεται σαν θέμα με την δυνατότητα των Παλαιστινίων να επενδύσουν Φερρυπίν στον τομέα Γ και να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχή υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προς τον Παλαιστινιακό λαό είμαι θα ευγνώμονες για την υποστήριξη της ε, αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Παλαιστίνη και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Σαλάμε και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Ρόμπερτ ε, Βάλετ, ειδικό απεσταλμένο ε, του διαχειριστή του προγράμματο του LTP για παροχή βόδια στον Παλαιστινιακό λαό να μα ενημερώσει για το πλαίσιο αθεκτικό της Παλαιστίνης. Είπα και προηγουμένω είναι η πρώτη φορά που αυτό το πλαίσιο αθεκτικότητα παρουσιάζεται σαν ένα από τα ευρωπαϊκά όργανα. Και να πω ότι ε, με τη συζήτησή μα και εμείς ε, θα συμβάλλουμε στην τελική διαμόρφωση του πλαισίου αυτού. Ο λόγο σε εσάς, κύριε Ροπέρτο Βάλετ. Seven minutes. Πέντε λεπτά. Είμαι Ιταλός. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αγαπητέ Πρόεδρε, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και Παλαιστίνης, Κύριε Σιλικιώτη, Αναπληρώτρη ε, επικεφαλής, κυρία Μάργαρετ Άουκεν, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμη καλεσμένη εξοχότητα κύριε Πρέσβη ε, της Παλαιστίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, διακεκριμένα μέλη του γραφείου σας. Δόκτωρ Στεφάν Σαλαμέ, ε, σύμβουλε του Πρωθυπουργού της Παλαιστίνης. Κύριε Έμαρσου Φάτεν, Διευθυντή του Trust Fund στην Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάδελφοι παριστάμενοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, εσάς και όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις Κοινοβουλίου με την Παλαιστίνη, για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθύνω το λόγο ε, στην ε, ομάδα σας και να ανταλλάξουμε υπόψη, απόψεις για την ανθεκτικότητα ή αντοχή των Παλαιστινίων και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει αυτή να ενισχυθεί σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Το Νοέμβριο του 2016, όπως είπε ήδη ο Δόκτωρ Σαλαμέ, η πρώτη διάσκεψη ανθεκτικότητας των Παλαιστινίων έλαβε χώρα στο Αμάν. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε με ειλικρίνεια ε, με ανοιχτό τρόπο τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται για τη στήριξη των Παλαιστινίων σε γενικές γραμμές. Πάρα πολλοί πόροι μαζικά ε, μαζικές ποσότητες πόρων μπαίνουν στη Παλαιστίνη σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο ανθρωπιστικής ε, δράσης για παράδειγμα και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το πλαίσιο δεν αλλάζει απαραίτητος για το καλύτερο. Και σε κάθε περίπτωση η πολιτική αιρεσιμότητα, οι πολιτικές προϋποθέσεις και η επίτευξη αυτών αποτελούν χαρακτηριστικό σημείο αυτού του ευρύτερου πλαισίου και η επιτυχία ε, όλων αυτών. Έχουμε την Εθνική Ατζέντα Πολιτική στην Παλαιστίνη και μπορέσαμε να συμβάλλουμε στην ε, διατύπωση αυτής ως διεθνής κοινότητα και η ε, η ατζέντα αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα και στους στρατηγικούς στόχους της ε, ε, ε ανάπτυξης. Είναι προνόμιο αλλά και ευθύνη η στόχη αυτή για την Παλαιστινιακή κυβέρνηση και αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήξει κανέναν εταίρο. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στο Αμάν είδαμε ότι υπάρχει ισχυρή ανθεκτικότητα των Παλαιστινίων η οποία υπονομεύεται και διαβρώνεται μετά από 50 χρόνια κατοχής και αποκλεισμό ε, και εμπάρκο στη Λωρίδα της Γάζας και το καθεξής μετά τις, όλες αυτές τις γνωστές εξελίξεις και ε, τίθεται εν κινδύνο η ανθεκτικότητα των Παλαιστινίων και η συνοχή τους. Αυτή τη στιγμή η οικονομία της Παλαιστίνης ε, στην καλύτερη περίπτωση βρίσκεται σε τέλμα και αυτό μας ανησυχεί. Η ενεργεία των νέων Παλαιστινίων και η υποαπασχόλησή τους βρίσκεται σε αστρονομικά επίπεδα. Στη λωρίδα της Γάζας έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σχεδόν παντού στον κόσμο και υπάρχει απελπισία, όλο και μεγαλύτερη απελπισία, έλλειψη ελπίδας και απόγνωση στη νεολαία των Παλαιστινίων και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση του Ισραήλ, με το Υπουργείο Αμήνες και οφείλω να πω ότι το, ο Υπουργός Αμήνης του Ισραήλ, εξετάζοντας με πολύ πρακτικό τρόπο τις διαστάσεις της ασφαλείας και τις επιπτώσεις όλης αυτής στη λωρίδα της Γάζας και το καθεξής, εκφράζει τις ανησυχίες του στο βαθμό που δεν είναι βέβαιος ότι μπορεί να στηρίξει τη δράση μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε επιτόπου στη λωρίδα της Γάζας και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Οι Παλαιστίνοι γίνονται όλο και πιο κατακαιρματισμένοι με μεγαλύτερο σκεπτικισμό, έχουν απολέσει την πίστη τους στην εθνική ταυτότητα, στην κοινωνική συνοχή, στην ειρηνευτική διαδικασία. Εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την βοήθεια και έχουν όλο και λιγότερη αυτάρκεια. Είναι σαφές ότι κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή είναι η τέλεια συνταγή για ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια, απελπισία, απόγνωση και αποσταθεροποίηση. Είναι αδύρυτη ανάγκη να ε, επαναπροσδιορίσουμε αυτή τη στρατηγική, την αναπτυξιακή, τη στρατηγική βοήθειας. Θα πρέπει η Παλαιστίνη να, να κάνει την αυτοκριτική της, να κάνει ε, μελέτες, να σκεφτεί προς τα που θέλει να κινηθεί και μετά από 50 χρόνια ανθρωπιστικής βοήθειας οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί όμως, για να πάμε στην αναπτυξιακή βοήθεια, να υπάρξει ανάπτυξη και η Παλαιστίνη συνεχίζει να θεωρείται ως επικράτεια όπου υπάρχουν ανθρωπιστικές ανάγκες και ανθρωπιστικά επίγοντα και ε, έχουμε θέμα φυσικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά είναι όψεις του ίδιου νομίσματος και δυσκολεύουν την ικανότητα των Παλαιστινίων να ε, ε, εφαρμόσουν κατάλληλες αναπτυξιακές στρατηγικές που θα αποσοβήσουν και θα εξουδετερώσουν την σοβούσα κρίση. Άλλωστε, ε, χρειάζεται πολιτικό πλαίσιο, καλοήθη ηγεσία που θα είναι και η πηξίδα, ο μπούσουλας για μεγαλύτερο ανθρωπισμό και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαρματίσει για την πρόθεση όλων αυτών των στόχων. Ε, το να αντιμετωπίζουμε τα πολιτικώς επίγοντα ζητήματα που προκύπτουν από τις πολιτικές συγκρούσεις που έχουν χρονίσει. Αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντισταθούν στις εξωτερικές πιέσεις. Σίγουρα όλα αυτά προκαλούν καταστροφές. Η ευαλωτότητα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων πολιτικής, όχι μόνο εθνικών αλλά και διεθνών αποφάσεων θα πρέπει και η διεθνής κοινότητα να έχει ένα σωστό πλαίσιο ανάπτυξης ε, με σωστή χρηματοδότηση, με εργαλεία management, εργαλεία διοίκησης για να καλλιεργήσει μια ανάπτυξη με ανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα στις συνθήκες. Αυτό αναφέρθηκε στο σχέδιο δράση του 2013 για την ανθεκτικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα κρίσιμο εργαλείο θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να στηριχθεί η στρατηγική ανθεκτικότητα και η δράση που έχουμε αναλάβει επιτόπου ε, στην Παλαιστίνη. Η προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών ε, και γενικότερα ο ΙΕ, γιατί με αυτή την ομάδα συνεργαζόμαστε, ε, τονίζεται η σημασία της μεταρρύθμισης των συστημάτων να εντοπιστούν τα συστήματα που υπονομεύουν την αθεκτικότητα και να εξουδετερωθούν για να έχουμε μια θετική αλλαγή, να έχουμε λιγότερη εξάρτηση, υψηλή παραγωγικότητα και αυτοδιάθεση, αποφασιστικότητα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να διαχειριστούμε την κρίση σε συνθήκες ευαλωτότητας και υψηλής εξάρτησης, όπου τα εξωτερικά σοκ ε, μπορεί να ανοίξουν τους χώρους που είναι απαραίτητοι για να υπάρχει μεταμόρφωση της οικονομίας που θα συμπεριλάβει περισσότερους, που θα θέσει τα θεμέλια για πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, ένα ανανεωμένο, ένα αναδιατυπωμένο εναρμονισμένο, επαναξιολογημένο πλαίσιο και καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Βλέπω ότι ξεπερνώ τα πέντε λεπτά, δεν μπορώ όμως να τα επεκταθώ σε αυτά. Θα ήθελα όμως να δώσω κάποια παραδείγματα, εν συντομία, δύο πολύ πρακτικά παραδείγματα που θα αναδείξουν τι εννοώ. ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στον τομέα της μεταποίησης και των κατασκευών. Στη λωρίδα της Γάζας η βιομηχανική περιοχή έχει κατεδαφιστεί, έχει, έχει εξουδετερωθεί, εξαλειφθεί πλήρω και θα πρέπει να αποκατασταθεί. Υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί και υπάρχουν λύσεις για την καλύτερη ένταξη της Παλαιστινιακής οικονομίας στην περιφερειακή και παγκόσμια αγορά. Και έτσι θα, οι, νέοι, οι γυναίκες, τα νοικοκυριά, τα φτωχά θα αποκτήσουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Θα μειωθεί η ανθρωπιστική βοήθεια μόνο για να αυξηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια, να δοθούν κίνητρα για καινοτομία και για επενδύσεις. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που προκύπτει από το Παλαιστινιακό πείραμα του τι συμβαίνει όταν δίνεις δυνατότητες και ικανότητες στους νέους, στις γυναίκες, στα αυτοχάνικο νοικοκυριά. Όταν έχεις το empowerment δηλαδή Έχουμε προγράμματα ε, που εφαρμόζει το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης που στηρίζει ε, το UNDP, τα Ηνωμένα Έθνη και δίνουμε συμπληρωματική στήριξη για στρατηγικές εξόδου από την κρίση μέσω προγραμμάτων μεταφοράς ρευστού ε, και θέλουμε ε, έχει, ε, ε, θέλουμε να μεταμορφωθεί, να αλλάξει η κατάσταση για τα νοικοκυριά. Από 22.000 νοικοκυριά έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα για να πάνε σε μια κατάσταση ανεξαρτησίας και αυτάρκειας θα δώσουμε στήριξη, ουσιαστική στήριξη και σε άλλα φτωχά νοικοκυριά, δημιουργώντας ευκαιρίες για απασχόληση, δίδοντας ε, πάνω από 45.000 μόνιμες θέσεις εργασίας και όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση του Παλαιστινιακού ΑΕΠ, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ε, το να ενισχύσουμε την αθεκτικότητα των Παλαιστινίων, αυτό χρειάζεται να είμαστε μαζί να ε, μειωθεί και να ε, καταργηθεί ο φραγμός μεταξύ του ανθρωπιστικού σκέλους και του αναπτυξιακού σκέλους. Αντιθέτως, να ενωθούν αυτά τα, δύο. τα δύο. Έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά στην Κωνσταντινούπολη στη σχετική διάσκεψη. Η αθεκτικότητα είναι κρίσιμη σημασίας, ζωτικής σημασίας όλοι ξέρουμε σε πόσο βαθμό έχουν μειωθεί οι ζωτικές ροές για την Παλαιστίνη. Χρειάζονται επίσης και νέοι πόροι. Ρόλος σας στην, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να βοηθήσετε για να επιστρέψει αξιοπρέπεια στο λαό των Παλαιστινίων, να προχωρήσουν προς την ανάπτυξη και να έχουν την ανθεκτικότητα για να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες. Ευχαριστώ. Ε, ε, πήραμε μια παράταση 10 λεπτών από την Ζερμινή. Ε, γι' αυτό θέλω να ζητήσω από τα μέλη να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Έχουμε στη διάθεσή μα ε, 5 λεπτά μόνο. Ε, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ε, θα θέσουμε ένα λεπτό και για να μπορούν να έχουν και τον χρόνο να απαντήσουν. Η Μαρτίνα. Μαρτίνα. Okay, I'll be very... Θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτη φορά που άκουσα για το πλαίσιο ανθεκτικότητας, όπως περιγράφει σήμερα. Και πρέπει να πω όταν ε, άκουγα την περιγραφή αυτού, θεωρούσα ότι ήταν περισσότερο ανθεκτικότητα προς επιβίωση. Ανεξάρτητα από αυτό που το περιγράψατε, δηλαδή ανθεκτικότητα για απελευθέρωση. Ίσως πρέπει να αποφασίσετε ποιος από τους δύο πάντως μια απάντηση πάνω σε αυτό. Δεν είμαι σίγουρη. Το θέτω σαν ερώτημα. Εγώ υποστηρίζω τη λύση των δύο κρατών και είμαι πολύ καλός φίλος του Παλαιστινιακού λαού και θέλω να δω κάθε κράτος μέλος να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο ανθεκτικότητας όσον αφορά τους νέους που χάνουν την πίστη τους στην ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό που είπατε, τη δυνατότητα να δημιουργηθεί βία, να υπάρξει απελπισία. Αν αισθάνονται ως απελπισμένοι αισθάνονται αν αισθανόμαστε εμεί απελπισμένοι, φαντάζομαι πώ πρέπει να αισθάνεται μια γενιά ανθρώπων που το ζει αυτό. Και πώ η ανθεκτικότητα που περιγράφεται έναντι των καταστραφών κατεδαφίσεων, όλα αυτά που αναφέρατε, ότι 40% της γης κατέχεται κλπ. Πώς το αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι. Λόγω σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Αναμφισβήτητα θα υποστηρίξουμε όσο μπορούμε στις προσπάθειές σας. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Κάποια θεσμικά όργανα πρέπει να κινηθούν περισσότερο από άλλη. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να αλλάξει τον τρόπο εργασίας της θα πρέπει να συζητήσουν το Ισραήλ. Είναι καλό να αντιμετωπίζεται έτσι οι Ισραηλινοί. Όχι θα μας πούν. Δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πάντα, να συμπεριλαμβάνουμε πάντα το Ισραήλ στα όσα κάνουμε. Να τους καλούμε να λογοδοτούν βέβαια. Τι χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα. Να, να στείλουμε μήνυμα ελπίδας να σχετίσουμε τις δράσεις μας με κάτι που μπορούμε να πετύχουμε τόπου. Είναι μακροπρόθεσμη η προπτική, συμφωνώ. Πρέπει να ζητήσουμε κάτι να γίνει. Να πω στην υπηρεσία της εξωτερικής δράσης ότι πολλά πράγματα υπάρχουν, υφίστανται. Δεν χρειάζεται να θεσπίσουμε νέο νόμο, υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει κάτι να υλοποιηθεί όμως. Τέλος, να πω κάτι άλλο. Είναι επικίνδυνο εμείς να λέμε ότι έχουμε καθυστερήσει, ότι είναι πολύ αργά. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Διότι αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί επιτόπου ο κατακτητής. Δεν πρέπει να μιλάμε εμείς έτσι. Μιλάμε για τα σύνορα του 67, επιμένουμε στα σύνορα του 67, ανεξάρτητα από αυτά που λέει το Ισραήλ. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι, οι βέβαια. Η γλώσσα αυτή, η διατύπωση δεν χρησιμοποιείται από εμά ότι είναι πολύ αργά. Μπορεί να είναι η πραγματικότητα αυτή αλλά εμείς πρέπει να πιέζουμε. Κάτι πρέπει όμως να γίνει. Πρέπει να αλλάξουμε τα προγράμματά μας και τον τρόπο εργασίας μας. Συμφωνώ. Ευχαριστώ Μαρκάλη. Ε, ήθελα και εγώ μόνο πολύ σύντομα κάποιες συμπροματικές ερωτήσεις. Το ένα είναι πώς συμπληρώνει το έργο του UNDP το πρόγραμμα εθνικής πολιτικής. Και το δεύτερο πώς ε, καταφέρνουμε να εμπλέκονται κοινότητες και ο ιδιωτικό τομέας ε, στην Παλαιστίνη σε αυτήν τη διαδικασία. Και να σας παρακαλέσω να είστε πολύ σύντομοι στις απαντήσεις σας. Thank you. Um, when we started... Όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας επ' αυτού, το Παλαιστινιακό Εθνικό Θεματολόγιο, την ατζέντα για την περίοδο 2017-2022. Πρώτα απ' όλα, είδαμε τι κάναμε πριν. Τι πήγε σωστά, τι πήγε στραβά. Το παρελθόν αναπτυξιακό σχέδιο της Παλαιστίνης υπέθεται ότι η Παλαιστίνη είναι ανεξάρτητη. Και σχεδιάσαμε προγραμματισμό βάσει ανεξαρτήτου κράτους. Αυτή τη φορά Προφανώς ανακαλύψαμε ότι τα πρώτερα σχέδιά μας δεν εδράζονται επί της πραγματικότητας. Αυτό, το τωρινό, το εξετάσαν πάλι σκοπιά. Τι χρειάζεται περισσότερο ο λαός μας. Πέρα από την απελευθέρωση, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ενότητα, αυτή είναι η πολιτική στόχη, ο λαός μας χρειαζόταν βασικές υπηρεσίες για να μπορεί ο λαός να σταθεί στα πόδια του και να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Παραδείγματο χάρη, είδαμε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή Γ. και γι' αυτό στην ατζέντα μας εστιαζόμαστε κατά πολύ επί ανθεκτικότητα, εστιαζόμενοι επί Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περιοχής Γ και Γάζας και μπορώ να σα δώσω και ένα απλό παράδειγμα. Αναφερθήκατε στο ΕΛΑΛΧΜΑΡ, αλλά υπάρχουν 46 κοινότητες Βεδουίνων σε στρατηγικές τοποθεσίες γύρω από την Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ καθημερινά απειλεί τις κοινότητες με καταναγκαστική ε, έξωση. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Παλαιστίνοι πριν ζητήσουμε τη στήριξη της κοινότητας. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτή η εθνική ατζέντα πολιτικής ασχολείται με τις πραγματικές συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες του Παλαιστινιακού λαού γνωρίζουμε ότι πρέπει να δώσουμε στις κοινότητες αυτές τις βασικές υπηρεσίες, να τους δώσουμε ελπίδα, να τους δώσουμε δουλειές, να τις προστατεύσουμε στο βαθμό του δυνατού. Αλλά ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι τελούν υποκατοχή και όπως είπατε, κυρία Άουκεν, Επίσης απαιτείται τεράστια πίεση από τη διεθνή κοινότητα ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα ανθεκτικότητας, να τεθεί τέρμα στην κατοχή και να δημιουργηθεί το Παλαιστινιακό κράτος. Ας δούμε και πιο δίκαιο και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παλαιστίνη. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τον κοινό προγραμματισμό όπως αποκαλείται και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διότι προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά συντόνισε σε τεράστιο βαθμό τις προσπάθειες μαζί μας για την κατάρτιση της ατζέντα εθνικής πολιτικής. Έχουμε μια καλή αφετηρία λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τον κοινό προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ενώση για την υποστήριξη της Παλαιστινιακής αντεκτικότητας. Υπάρχουν προγράμματα που φροντίζουν την υποστήριξη της παιδείας στην Παλαιστίνη και του συστήματος υγείας, κυρίως σε περιθωριοποιημένες κοινότητες. Έχουμε προγράμματα τα οποία θα καταπολεμήσουν την πολιτική κατεδαφίσεων του Ισραήλ και θα προβλέπεται πρόγραμμα ανοικοδομήσεων. Έχουμε προγράμματα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των κοινοτήτων των Βεδουίνων και επίσης προβλέπουμε και προγράμματα για την ενέργεια, για το νερό, για τις Παλαιστινιακές κοινότητες στην περιοχή Γάμα, στη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κυρίως για τα προγράμματα στέγασης και τα προγράμματα εκπαίδευση Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στον συνάδελφό μου τον Ρομπέρτο. Ένα λεπτό σου αρκεί νομίζω, Ρομπέρτο. Εντάξει, ένα λεπτό λέει ο Ρομπέρτο. Το ερώτημά σας, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πώς το UNDP ε, συμπληρώνει τα όσα κάνει η Παλαιστίνη. Πρώτα απ' όλα ενταζόμεθα στο θεματολόγιο το εθνικό. Αυτό κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. δεν θέλουμε, δεν θεσπίζουμε στρατηγικές απομονωμένα. Σε UNDP κινούμεθα στο πλαίσιο της ομάδας του ΟΗΕ, η συγκεκριμένη χώρα, αλλά είμαστε εντός της UNDAP. Στο πλαίσιο αναπτυξικής βοήθειας του ΟΗΕ. έχουμε πάνω από 20 φορείς επιτόπου, άρα απαιτείται συντονισμό και η UNDP μόλις πέρσι ανοικοδόμησε μέσω υποστήριξη αυτοβοήθειας των Παλαιστινίων στη Γάζα πάνω από 13.000 σπίτια ανοικοδομήθηκαν που είχαν καταστραφεί σαν αποτέλεσμα συγκρούσεων. Εργαδόμεθα επικά του δικαίου και προσβάσα στη δικαιοσύνη, βασικά ανοικοδομώντας υποδομές όπως το σύστημα της δικαιοσύνης, τα δικαστήρια, Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όλο τον τομέα της δικαιοσύνης και το σχετικό σύστημα σε συντονισμό με διάφορους φορείς όπως UNICEF και USCR, η Πατερμοστία. Εργαζόμαστε με τους τρεις κλάδους της δικαιοσύνης στην Παλαιστίνη και στη Γάζα με υποστήριξη από Κατάρ κινούμεθα για στήριξη της παιδείας, για στήριξη σχολείων και συνεργαζόμαστε μόνο τα πανεπιστήμια. Κινούμεθα επί μεταρρυθμίσεως ε, του τομέα του δημοσίου και ολοκλήρωση του δημόσιου τομέα και της παροχής υπηρεσιών προς πολίτες. Είναι δύσκολος δρόμος. Απαιτείται και κάποια πολιτική απόφαση στον τομέα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βάλε και τον Δόκτωρ Σαλάμε για την ε, σημαντική συμβολή του. Ε, αυτό που θέλω να βεβαιώσω, αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί. Νομίζω είναι ένα τομέα που και εμείς ως αντιπροσωπεία ε, με την Παλαιστίνη πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο ε, και πρέπει να πω στην εκπρόσωπο της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης δεν ακούγεται μόνο κριτική για την υπηρεσία εδώ. Άκουσαμε πολύ καλά λόγια από τον δόκτωρα Σαλάμε για τη βοήθεια και το γνωρίζουμε και εμείς και πολλές φορές είπαμε για τη βοήθεια που δίνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης στην Παλαιστίνη. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και τη συμβολή σας στη συζήτηση. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς ε, για την σημαντική συμβολή τους ώστε να διεξαχθούν ομαλά οι εργασίες ε, της συνεδρίας μας. Η επόμενη συνεδρία ενδεικτικά είναι 8 Μαΐου. Ε, η συνάντηση αυτή, η συνεδρία αυτή θα γίνει με τη συμμετοχή του βουλευτή του Ισραηλινού Κοινοβουλίου του Αχμετίπου από την κοινή λίστα στο γραφείο της αντιπροσωπείας έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε αυτή η συνάντηση να γίνει από κοινού αν είναι δυνατόν με την αντιπροσωπεία με το Ισραήλ. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Thank you very much. Thank you very much. Sorry for the short because you have this issue about the prisoners. It was needed to discuss that because it's, uh, sometimes you have ethics. it's, it's, it's a priority.